την φωτογραφία αυτή που δείχνουν ότι υπάρχει μια κοινή δράση όλων των θεσμικών οργάνων με την παρουσία της φωτογραφία. Ωραία λέει Σας ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα κυρίε και κύριοι στις ψηφοφορίες. Έχουμε στην αρχή την έκθεση Κάου για την άρση της ε, ε, ασυλίας του κυρίου Έρενχάουζερ. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές έχει ούτως αποφασιστεί. Περνάμε τώρα στον προϋπολογισμό 2013. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λαβία, στον εισηγητή. Παρακαλώ κύριε Λαβία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως κάθε χρόνο, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας του προϋπολογισμού, υπάρχουν ορισμένες τεχνικές προσαρμογές που θα πρέπει να ψηφίσουμε. Καταρχήν, κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι τα στοιχεία για το λεγόμενο το έγγραφο 6. Υπάρχουν ορισμένε τροπολογίε και μετά υπάρχουν ορισμένα στοιχεία για τι προπαρασκευαστικέ δράσει που θα πρέπει να, να ψηφίσουμε. Υπάρχει το σχέδιο για του δείκτε για, για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα ανδρών και γυναικών στην τοπική ε, ζωή. Έχει εγκριθεί στο, στην κατηγορία 3 και όχι στην 1α. Επίσης, η προπαρασκευαστική δράση για την κατανάλωση οπροκυπευτικών είναι στην, στο 2, κατηγορία 2 και όχι 3β. Το σχέδιο για τα συστήματα υγειονομικής αυτοϋποστήριξης είναι 1 εκατομμύριο ευρώ και όχι 100.000. Η προπαρασκευαστική δράση για τις κλιματικές ε, ενέργειες και την καιροτομία είναι 2 εκατομμύρια λιγότερα από το σχέδιο προϋπολογισμού η δράση προπαρασκευαστική για το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα έχει μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο σε σχέση με το σχέδιο προπολογισμού και στι υποχρεώσει και στι πληρωμέ. Επίση, θέλω να αναφέρω ότι σχέση στη θέση του Κοινοβουλίου δεν λαμβάνει υπόψη την διαρθωτική επιστολή 1-2013 που ενεκρίθη στι 19 Οκτωβρίου από την Κομισιόν και η οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί μετά μέσα στη διαδικασία συνδιαλλαγή. Θα ήθελα τέλο να κάνω μια έκκληση σε όλου η Ένωση και η συνοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πιο σημαντικέ από ποτέ για τον προπολογισμό του 2013. Θα έχουμε μια δύσκολη διαδικασία συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο, η οποία που το Συμβούλιο δεν δείχνει ότι θέλει να απελευθερώσει του απαραίτητου πόρου. Χρειαζόμαστε μια στεναρή θέση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι ψηφοφορίε για να δείξει ότι είμαστε έτοιμοι ενωμένοι να αποδειθούμε σε αυτό το αγώνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Λαδία, Πράγματι θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν πιο ενωμένοι να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα οποία πρότεινε ο κύριος Λαβία ήδη, τα οποία έχετε ε, λάβει υπόψη, να ψηφίσουμε για όλα αυτά τα σημεία που αναφέρει ο κ. Λαβία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές με μεγάλη πλειοψηφία έχουν γίνει δεκτές. Περνάμε στο μπλοκ 1. Ψήφι υπέρ. Το μπλοκ 1. Ψήφι υπέρ. Όχι, όχι, συγγνώμη. Το μπλοκ 1, από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, γίνεται δεκτό. 901 ψήφι υπέρ. 891. Απορρίπτεται. 791 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο για την 791. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. 2.72 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.51 ψήφι υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Δεκτή. 878 εκπίπτει. 206 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 774 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 200 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. Κύριε ε, Ντες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν λειτουργεί το σύστημά μου για την ψηφοφορία, πρέπει να σας πω δυστυχώς. Ένας τεχνικός πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Άμα βγάλετε την κάρτα και την ξαναβάλετε, πολλές φορές λειτουργεί το σύστημα πάλι. Ε, δεν, δεν λειτουργεί ακόμα. Ε, εντάξει. 963 εκπίπτει. Ερχόμαι στην τροπολογία 964 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, όλες, πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην ψηφοφορία 965 σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση. Αρχίζουμε την ψηφοφορία στο πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Και το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 966. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 1200. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 1200 ψήφοι υπέρ. Επαναλαμβάνω. Κατά. Είτε δεκτή. Σαφώς. Άμα θέλετε κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Είναι σαφές όμως το αποτέλεσμα. 1200. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Είτε δεκτή. 116 εκπίπτει. 762 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 εκπίπτει. Ως συνέπεια. Ονομαστική κλίση 899. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. 1162 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ως αποτέλεσμα εκπίπτει 190. Ερχόμαστε στη 280. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απολύτω. 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μπλοκ 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μπλοκ 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33. Υπέρ κατά απόχες δεκτή 29 υπέρ κατά απόχες δεκτή 9 9.98 Α, εκπίπτει γιατί ανακρίθησαν οι προηγούμενες 11.48 με ονομαστική κλίση άρχεται την ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται επομένω η 876 εκπίπτει 1005 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες 754 και 997 ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Αλλά δεν έχει φτάσει την ειδική πλειοψηφία, επομένως δεν εγκρίνονται. 1002. Ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 992 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπλοκ 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> Δεκτή. Δεκτό. Τροπολογία 977 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 298 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Εγκπίπτει η 978 ως ε, αποτέλεσμα. 793 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται εκπίπτει η 979 ως αποτέλεσμα τροπολογία 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 891 εκπίπτει ως αποτέλεσμα 1147 με ονομαστική κλίση, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε η επόμενη 892 εκπίπτει. 808 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έτσι 741. Όχι. Φαίνεται ότι έχει καταπέσει μεν ε, το αριθμητικό, αλλά πρέπει τις εξηγήσεις να τις ψηφίσουμε. Υπέρ παρακαλώ, τις ψηφίζουμε. Οι ομάδες νομίζω είναι και αυτές σου, σε σύγχυση όσο και εμείς. Παρακαλώ, κατά Απορρίπτεται. 781 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11.52 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έτσι η 893 καταπίπτει. Στο 5 τώρα υπέρ κατά. Αποχές εγκρινεται στο 6, μπλοκ 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 274 υπέρ κατά άποχες απερίφθη 1018 1018 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ε, ε, 1240 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται παρακαλώ. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 939 καταπίπτει. 1241 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1192 πάλι δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ας το επαληθεύσουμε. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία δεύτερο τμήμα της 1192. Υψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 262, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Ναι, έχετε δίκιο. 1194 ονομαστική. 1194 πάλι ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. 220 και 1020 καταπίπτουν. 1195 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και έτσι οι τροπολογίες 221 και 1021 καταπίπτουν. Τροπολογία 432. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 222 και 1022 καταπίπτουν. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 947 καταπίπτη 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 948 καταπίπτει ως εκ τούτου ή 244 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται παρακαλώ εψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Και έτσι καταπίπτει 935, 245 υπέρ. Με συγχωρείτε, ονομαστική ψηφοφορία λέει ο πρόεδρος, άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και καταπίπτει 932. 1243 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται και καταπίπτουν οι 226, 1024 και 1045 και τώρα πάμε στην 1255 παρακαλώ υπέρ, 1245 υπέρ, ε, ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. εγκρίνεται και καταπίπτουν οι ακόλουθες για να περάσουμε στην 1246 πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι, πέρας. εγκρίνεται και η επόμενη ακριβώς καταπίπτει η 247 παρακαλώ ψηφίζουμε κατά αποχές εγκρίνεται αλλά αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας ψηλά δεν μπορώ να σας βλέπω και να καταλάβω ότι ψηφίζετε μπορεί να θέλετε να κρατήσετε το κεφάλι σας πάνω στο χέρι σας καταπίπτει λοιπόν η 275 και πάμε στην 1196 παρακαλώ ονομαστικά άρχιτη ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται και καταπίπτουν οι επόμενες ε, τροπολογίες και πάμε στην ομάδα 7, μπλοκ 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1258 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται παρακαλώ εψήφισαν όλοι Πέρασε. εγκρίνεται Ακολουθούν οι επόμενε τροπολογίες και πάμε στο μπλοκ 8, ομάδα τροπολογιών υπαριθμών 8, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 1263 τώρα ονομαστική ψηφοφορία υπέρ μάλλον συγγνώμη λέει ο πρόεδρος άρχεται η ψηφοφορία είναι λίγο αργά τα μηχανήματά μας σήμερα εψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορία σου.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 Παρακαλώ κύριε Μαυρογέννη. Για λόγους διαδικαστικούς, κύριε Κονπεντήτη, είναι υποχρεωτικό να δώσω το λόγο. Κύριε Μαυρογιάννη. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου το σχέδιο προπολογισμού για το 2013. Πράγματι, συνεπώς, υπό την ιδιότητά μου ως Προεδρεύων του Συμβουλίου, σύμφωνο να συγκαλέσει την Επιτροπή Συνδιαλλαγής ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 γάμα της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαβία, θέλατε κάτι να πείτε σε αυτό. Παρακαλώ. Αφήσαμε μια τροπολογία, τι ψηφίσαμε, την 262 του κεφαλαίου 4, της κατηγορίας 4, δεν ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία. Α, κατέπεσε. Καλώς. Okay. So... Εντάξει λοιπόν, ευχαριστώ. Τώρα, να δούμε την έκθεση Λαβία Βόν. Τα τμήματα για τον προϋπολογισμό παρακαλώ. Αν δεν θέλει κανείς το λόγο, ξεκινάμε με την πρώτη 18 υπέρ, με την παράγραφο 18 υπέρ, κατά, αποχές. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 44 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 45 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 21 για το 18 για την παράρφη 18 αρχιψηφορεί ονομαστικά παρακαλώ εψήφισαν όλοι πέρας απερίφθη 36 τώρα παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές. Απεριφθεί στο αρχικό κείμενο πάλι. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και στα δύο τμήματα και τώρα στο 22, όχι, τροπολογία 22, γάμα, 22C, e ECR, α, D, 22D της ECR, υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Το 19 τώρα, υπέρ, υπεράχος 19, κατά, αποχές απερίφθη. Τροπολογία υπαριθμών 1, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Τώρα στην δεύτερη τροπολογία, με ονομαστική ψηφοφορία και πάλι, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι, πέρας. Απερίφθη. Τρία, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μα, το, σας ρωτάω να σηκώνετε και τα χέρια. Υπέρ της 38. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε όμως. Δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. 38. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απερίφθη. Τροπολογία 4, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Σαράντα τροπολογία 48 υπέρ, κατά αποχές, απερίφθη. Η τροπολογία 5 ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 8 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Υψήφισαν όλοι. Πέρασε. απερίφθη. Η τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 41 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ωραία, ε, επαλήθευση, Άρχιτε ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Α, Απερίφθη προφανώ. 15, τροπολογία 15, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 16. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. πέρασε. Απερίφθη 26 και πάλι ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ, άρχεται. Και ψήφισαν όλοι, πέρας. Απερίφθη 27 υπέρ, κατά. Αποχές, απερίφθη 28 ονομαστικά, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας. Πέρας. Απερίφθη. 29. Ονομαστικά και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο τώρα στο, στην παράγραφο 86. Υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αρχικό τμήμα, τμήμα ε, κείμενο της 88 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία ονομαστική ψήφισαν όλοι Πέρασε. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα και πάλι ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο της 89 παρακαλώ, σε διατμήμα το πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά και πάλι, άρχεται. Ψήφισαν όλοι, Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 90 πάλι ονομαστικά. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλώς, αν θέλετε. Τροπολογία 11, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο. Στην παράγραφο 91 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 31, δύο τμήματα. Πρώτο παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 17 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 34 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι ορατό το αποτέλεσμα, επομένως κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα το ψήφισμα το ψηφίζουμε συνολικά με ονομαστική ψηφοφορία, Άρχη ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στους εισηγητές. Και τώρα έχουμε την έκθεση των κυρίων Μπέγκε και Κάλφιν. Τροπολογία 47, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται παρακαλώ. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 61, στην πρώτη παράγραφη, υπέρ, κατά, άποχες, απερίφθη. 39 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Μπορούμε να ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες της ΓΟΕ 49-64 ομού, εάν δεν έχετε αντίρρηση και αν δεν έχει πάνω από αντίρρηση η να τις ψηφίσουμε ομού, συμφωνείτε. Έχει κανείς αντίρρηση να ψηφίσουμε ομού τις τροπολογίες αυτές. Ψηφίζουμε λοιπόν 49, 50, 51, 52, 53, 63 63, 64, en παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Και πάμε στην τροπολογία 40, ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ, έρχεται. ψήφισαν όλοι, πέρας. Απερίφθη. 41 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Όχι, δεν το κάνω πια. Το κάναμε με το EFD μια φορά, δεν θα το ξανακάνουμε. 42 παρακαλώ ονομαστικά ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 43. Ονομαστικά. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τροπολογία 5 ονομαστικά άρχιτε ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 44 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας Απερίφθη. Η 66 τώρα υπέρ. Κατά. Εποχές. Απερίφθη. 6. Τροπολογία 6. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. 6D. Απερίφθη. 7D. Ονομαστικά. Άρχιτε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 8D. Ονομαστικά. άρχιτε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 9D. Ονομαστικά. άρχιτε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 45 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 67 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 10 ονομαστική ψηφοφορία υπέρ. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Εάν ε, δέχεται η ΕΦΔ μπορούμε να ψηφίσουμε την 11 η τη 12 η και τη 13 η ομού. Ένα λεπτό. Νέιου. Ναι λοιπόν, καλώς. Όχι, όχι. 11D ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. Δύο. ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 68 υπέρ. Όχι, προφανώς απερίφθη. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 56 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 72 υπέρ κατά αποχές απερίφθη το αρχικό κείμενο Ας επαληθεύσουμε την 72 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απερίφθη. Αρχικό κείμενο. Στο 72 πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 14 αντί ονομαστικά υπέρ Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απερίφθη 69 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 15D ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Απερίφθη. 16D. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν Πέρας. Πέρασε. Απερίφθη 17D. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Απερίφθη. 18. Δύο ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη, 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 19 αντί ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. απερίφθη. Η 20D επίσης ονομαστικά άρχεται. Πέρασε. Απερίφθη. Κύριε Λάμστορφ. Πρόεδρε, ψηφίσουμε πολλές τροπολογίες μίας μόνης ομάδας η οποία από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερα προσπαθεί να επιβάλλει αυστηρότατη τήρηση του κανονισμού. Θα έλεγα για τα πολύ σημαντικά θέματα των τροπολογιών αυτών να δοθεί η δυνατότητα να επανεξεταστεί από τις υπηρεσίες μας σε συνεργασία με την εν λόγω ομάδα το κατά πόσον είναι απαραίτητο πράγματι να γίνεται ονομαστική ψηφοφορία. 21 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Ατροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απερίφθη. Ερωτώ την ομάδα EFD εάν δέχεται την 22, 23, 24, 25, 26 και 46 να τις ψηφίσουμε on block. Κύριε Σπερώνη, εσείς είστε προεδρεύον της ομάδας. Ωραία, λοιπόν, ομού την ομάδα αυτή των τροπολογιών. Άρχεται η ψηφοφορία. Μα ούτε καν είστε μέλος της ομάδας αυτής εσείς. Τι λέτε, η ομάδα είπε ότι δέχεται ομού ψηφοφορία. Όχι, όχι, 22 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 23D. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 25D. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 26 άρχεται. Πέρας απερίφθη 46 άρχεται πέρας Απερίφθει. 50 στο, στο αρχικό κείμενο ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία εψήφισαν όλοι πέρας ψήφισαν όλοι πέρας Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 27 αντί υπέρ. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 28 αντί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη 29 αντί άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη 30 D άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη 31 D άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απερίφθη 32D άρχεται ψηφοφορία πέρας απερίφθη 75 άρχεται η ψηφοφορία κατά αποχές εγκρίνεται 33D ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρας Απερίφθη. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 34-2 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 35D ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 70 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 36D ονομαστική ψηφοφορία άρχιτη ψηφοφορία πέρας απερίφθη 37D άρχεται πέρας απερίφθη 71 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 80 38D έρχεται η ψηφοφορία πέρας απερίφθη. Εβδομήντα 76, 76 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 80 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται Τέσσερα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας απερίφθη τώρα πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται και συγχαρητήρια στους κυρίους Μπέγκε και Κάλφιν. Νομίζω ότι μετά τις πλειοψηφίες οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ ξεκάθαρες εν των διαπραγματεύσεων που πρόκειται να ξεκινήσουμε τη συνδιαλλαγή και αυτό ενισχύει σημαντικά τη θέση μου. Σε ευχαριστώ θερμά για την ευρύτατη αυτή υποστήριξη. Και τώρα έχουμε την έκθεση του άρθρου 138 του κυρίου Ντεχάν, μία ψηφοφορία με ονομαστική, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. Και τώρα πάμε στην έκθεση της κυρίας Γκρέσλε και Ριβελίνη για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό και οι δύο θέλουν το λόγο εν συντομία πριν από την ψηφοφορία. Πρώτη κυρία Γκρέσλε παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα ψηφίστε ένα ενοποιημένο, ενοποιημένο κείμενο με ένα, με μία ψηφοφορία και για τις ε, επεξηγήσεις αλλά και για μία ε, δήλωση που θα πρέπει να σας διαβάσω. τα, 50, τα 85,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ε, επέστρεψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Βέλγιο έχουν ε, δεσμευθεί με βάση το άρθρο 18 για την χρήση σε συγκεκριμένου σκοπούς. Αυτή είναι η διατύπωση την οποία έχουμε συμπεριλάβει τώρα ως επεξήγηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν ε, μέρος σε αυτή την προσπάθεια και μας βοήθησαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ριβελίνη τώρα. Πολύ πιο σύντομα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σήμερα εγκρίνουμε ένα νέο κανονισμό, πιο σύγχρονο, πιο απλό για τη διαχείριση των πόρων που έχει πιο αποτελεσματικέ διατάξει για να αντιμετωπίσει και να νικήσει τι προκλήσει τη παρούση κρίσεω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλου. Ευχαριστώ κύριε Ριβελίνη. Το κείμενο του κανονισμού ως ένα με μία ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται και τώρα Η πρόταση όπως τροποποιήθηκε σε μία ενιαία ψηφοφορία τώρα ψηφίσουμε παρακαλώ υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Πρόταση νομοθετικού ε, ψηφίσματος δυνάμει του πρώτου άρθρου με την προηγούμενη διαδικασία. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται για το νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε επεξηγήσεις ψήφου. Με τον κύριο Φόξ πρώτο. Έκθεση Λαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα αντιμετωπίζουμε την πολύ άσχημη οικονομική κληρονομιά της προηγούμενης εργατικής κυβέρνησης. Χρειάστηκε να αυξήσουμε τους φόρους και να μειώσουμε τις δαπάνες. Καταψήφισα τον σημερινό προπολογισμό γιατί προτείνει αύξηση στις δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 6,8%. Το να ζητάει τέτοια μεγάλη αύξηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιαδήποτε αύξηση, είναι παράλογο και ε, δείχνει έλλειψη ευαισθησίας. Θα απομακρύνει του ψηφοφόρου του Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ένωση.